μεταξύ που είναι η δήλωση τη Επιτροπή, Διαφάνεια και έλεγχο Κλινικών Δοκιμών. Και τώρα δίνω το λόγο και πάλι στον Επίτροπο, τον κύριο Αντρουκάητη. Έχετε το λόγο εκ μέρου τη Επιτροπή. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, θα ήθελα να εκφράσω την ε, συμπαθιά μου και τα συλληπιτήριά μου για τα θύματα που ε, κατέληξαν κατά τις κλινικές δοκιμές στη Γαλλία και στις οικογένειές τους. Να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου. Πιστεύω ότι οι γαλλικές αρχές πήραν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν ε, την κατάσταση και ότι βάζουν τη δυνατά τους για να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη και είμαι προσωπικά σε στενή επαφή με το αρχικό με το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας ε, για να παρακολουθώ τις νέες εξελίξεις στην έρευνα. Είναι σημαντικό όλοι να αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής πριν να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Οι κλινικές δοκιμές είναι ουσιαστικές για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και για την βελτίωση των θεραπείων που χρησιμοποιούν ήδη εγκεκριμένα φάρμακα. Οι κλινικές δοκιμές προσφέρουν ελπίδα σε ασθενείς που υποφέρουν από σπάνιες νόσους ε, σε ε, τομείς όπως η παιδιατρική ογκολογία. Υπάρχουν σύνδεσμοι μεταξύ της συμμετοχής σε κλινικές δοκιμές ε, και του προσδόκιμου ζωής των ασθενών δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένο κίνδυνος συνδέεται με οποιαδήποτε κλινική δοκιμή. Οι κλινικές έρευνες είναι ένα τομέα όπου έχει ηγετική θέση η Ευρώπη και συχνά ευρωπαϊκό, στον ευρωπαϊκό χώρο γίνονται οι πιο καινοτόμε ε, θεραπείες και αυτό είναι ο κύριο στόχος ε, του νομοθεσία μας. Ε, θα πρέπει να είναι δυνατό να ξέρουμε ποιες κλινικές δοκιμές συνεχίζονται, πού γίνονται, από ποιον και ποια είναι τα κριτήρια του. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες διατίθενται ήδη βάσει του υφιστάμενου μητρώου κλινικών δοκιμών που ε, είναι υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Επιπρόσθετα, όταν μία κλινική δοκιμή έχει ολοκληρωθεί, το αποτέλεσμα της θετικό ερνητικό θα πρέπει να δημοσιεύεται. Επίσης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμακών, ο ΕΜΑ, έχει ακολουθήσει μία πολιτική να υποβάλλεται μία ε, έκθεση ως τμήμα της χορήγησης ε, άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων. Έτσι λοιπόν πραγματικά η Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη θέση σε σχέση με τα δεδομένα. Όμως ε, ο νέος κανονισμός θα φέρει μία πραγματική βελτίωση στη διαφάνεια. Όλες οι πληροφορίες στις κλινικές δοκιμές που έχουν τα κράτη-μέλη στην Ευρώπη θα αποθηκεύονται σε μια νέα βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι από τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ορισμένες εξαιρέσεις, το όλο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι δημόσιο. Επίσης, ε, σε περιπτώσεις ε, δημοσίου συμφέροντος, όλες οι πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες δοκιμές θα δημοσιεύονται αμέσως. Ε, η Βάσει αυτή των δεδομένων αναπτύσσεται από την ΕΜΑ και αυτό το εργαλείο είναι ζωτικό για να λειτουργεί σωστά ο νέος κανονισμός. Θα βοηθήσει ταυτόχρονα να διαχειριζόμαστε τη ροή των πληροφοριών που αφορούν χιλιάδες κλινικές δοκιμές που υλοποιούνται καθημερινά στην Ευρώπη και σίγουρα αποτελεί ένα πολύπλοκο project πληροφορικής, κατανοώντας όλες τις τεχνικές προκλήσεις. Λυπάμαι που λέω ότι αυτό το σχέδιο έχει καθυστερήσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο Οργανισμό Φαρμάκων, τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα πρέπει να καταβάλουν πιο σκληρέ προσπάθειε έτσι ώστε να καταστεί λειτουργική βάση δεδομένων το συντομότερο για να υπάρξει πλήρη εφαρμογή του νέου κανονισμού. Τώρα δεν ε, υπάρχουν στοιχεία που να μας δείχνουν ότι η εφαρμοσιμότητα του νέου κανονισμού ε, θα είχε αποτρέψει τα γεγονότα στη Γαλλία. Είμαι σίγουρος ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα χρησιμοποιήσει του απαραίτητους τεχνικούς πόρους και η Κομισιόν θα το παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυ. Επίσης, καλό όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν ε, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, γιατί μερικές φορέ είναι δύσκολη η συνεργασία. Καλό τα κράτη-μέλη να ενδυναμώσουν ε, τη συνεργασία τους για αυτό το έργο και να κλείσω υπογραμμίζοντας εκ νέου τη σημασία τη αυξημένη διαφάνεια των κλινικών δοκιμών δοκιμών στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτευχθεί υπό το νέο κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές. Απευθύνω έκκληση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν εκ του συνεγγύς για να καταστεί εφαρμοστές ο κανονισμός το συντομότερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ο λόγος στους βουλευτές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Και Λίζ δεν είναι εδώ από ό,τι βλέπω. Ε, και χρότε. Δύο λεπτά. Τότε να μιλήσω εγώ για το ΕΛΚ. Όχι. Οι κλινικές ε, δοκιμές και, και τα περιστατικά στην ε, Γαλλία, στην ουσία, είναι μια καταστροφή. Πραγματικά θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τη συμπονιά μου στα θύματα. Παρ' όλα αυτά, αυτές αυτή η καταστροφή το 2006 στο Northwick μας έδειξε πώς πρέπει να γίνονται οι κλινικές δοκιμές. Αυτό ήταν σωστό. Υπήρξε μεγάλη ασφάλεια και ε, είχαμε ε, χιλιάδες ανθρώπους που έλαβαν μέρος στις κλινικές δοκιμές. Το πρόβλημα τώρα και το ζήτημα είναι η ενημέρωση. Να γνωρίζουν δηλαδή σε τι συμμετέχουν και ποια είναι η επίπτωση αυτή αυτών των περιστατικών στην εφαρμογή της νομοθεσίας που έχουμε αποφασίσει στο Κοινοβούλιο και με το, σε συνεργασία με το Συμβούλιο για τις κλινικές δοκιμές και τι πρέπει να περιμένουμε ως προς την βάση δεδομένων. Έχουμε πει ότι πρέπει να είμαστε διαφανείς, πρέπει να συζητούμε ανοιχτά και γι' αυτό υπάρχει μια βάση δεδομένων. Ε, θα περιμένουμε λοιπόν ότι θα εφαρμοστεί αυτή η βάση δεδομένων και θα είναι online. Επίσης πρέπει, θα πρέπει σε αυτή τη φάση 1 ε, για τους ασθενείς να προσέξουμε ε, πώς ακριβώς ε, θα προχωρούμε. Πρέπει η Κομισιόν να κάνει κάτι περισσότερο. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά την νομοθεσία μας ως προς τις έρευνες. Η ομάδα μου ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γι' αυτό και θα ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη συζήτηση για ένα θέμα που τόσο αφορά τον κόσμο, το κοινό. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένω να δω αν ε, ε, έλθει ο συνάδελφος Λίζε, αλλά μέχρι τότε η κυρία Ρης. κλινικές δοκιμές γνωρίζουν δημοσιότητα. Όσοι συμμετέχουν συμμετέχουν στην πρόοδο της ιατρικής. Μετά στην ΡΕΝ στις 10 Ιανουαρίου είχαμε αυτό το ατύχημα 10 ασθενείς εισήχθησαν στο νοσοκομείο ε, μεταξύ μιας ομάδας δηλαδή θελοντών σπάνιο περιστατικό αλλά πολύ σημαντικό. Και εγώ με τη σειρά μου επιτρέψτε μου να στείλω τη σκέψη μου στις οικογένειες των θυμάτων που παλεύουν ακόμη για την υγεία τους. Υπενθυμίζω ότι οι δοκιμές αυτές είναι βεβαίως απαραίτητες πριν την κυκλοφορία στην αγορά κάθε φαρμάκου. Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει πρωτοπόρο στις σχετικές έρευνες. Θυμίζω το Βέλγιο, στο Βέλγιο παράγονται παράγεται το 15% των ευρωπαϊκών φαρμάκων. Θέλουμε να παραμείνουμε στην πρωτοπορία. Δύο ερωτήσεις έχω προς τον Επίτροπο για την διαφάνεια. Κύριε Επίτροπε, είναι αλήθεια ότι η δημοσίευση όλων των αποτελεσμάτων των δοκιμών μετά από όλες αυτές τις διαπραγματεύσει. ότι η υποχρέωση αυτή λοιπόν δημοσιότητα αναβάλλεται και ισχύει ότι οι τάσει στα εργαστήρια στην Ευρώπη είναι να δημιουργούν παρέλες ομάδες ασθενών μεταξύ των οποίων η πρώτη λαμβάνει πολύ ψηλότερες δόσεις όπως έγινε και στη Ρέννα στο γνωστό ατύχημα λόγω ακριβώς των μεγαλύτερων δόσεων. Μήπως αυτό είναι αποτέλεσμα του εντονότερου ανταγωνισμού στον τομέα. Φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο αγώνας αυτό, ο ράλι, ο αγώνας δρόμου η την ε, επικύρωση των ε, δοκιμών δεν βοηθάει την υγεία των Ευρωπαίων. Πρόεδρος Χάζεκαμπ χωρίς μικρόφωνο Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ πριν κυκλοφορήσει ένα φάρμακο, πριν κάνει δοκιμές, το φάρμακο δοκιμάζεται σε ζώα. Σε ποντίκια, κουνέλια και ούτω καθεξής. Απαγορεύεται η χρήση πυθίκων στην Ευρώπη. Υπάρχει ένα θέμα ηθικής εδώ, όταν προκαλείται πόνος. Υπάρχει όμως και θέμα προβλεψιμότητες βεβαιότητε περί του κατά πόσο είναι ασφαλή φάρμακα αφού δοκιμαστούν σε ζώα. Ισχύει αυτό και του ανθρώπου. Φοβούμαι ότι θέτουμε, όπω είδαμε και στη Γαλλία, ανθρώπινε ζωέ σε κίνδυνο. Η ουσία αυτή, όπως είπε και ο Γάλλος υπουργό, είχε δοκιμαστεί ακόμα και σε χιμπατζίδες. τι όμω. Ερωτώ λοιπόν, Πώ είχε δοκιμαστεί η ουσία σε χιμπατζίδε παρά το ότι απαγορεύονται αυτέ οι δοκιμέ στην Ευρώπη. Και θα μπορέσουμε επιτέλου να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστα μοντέλα δοκιμών που να αφορούν του ανθρώπου, Πρόεδρο. Ένα μισή λεπτό, κύριε Ριβαζή. Κύριε Πρόεδρε, δεν αμφισβητώ την τιμιότητά σα. Να ξεχωρίσουμε όμω τα κριτήρια από τις δοκιμές τις ίδιες. Εγώ θέλω να πω, σαν αφορά τις κλινικές δοκιμές, ότι στις 17 Δεκεμβρίου του 2015 ένας άνθρωπος πέθανε στο πλαίσιο δοκιμών στο γνωστό νοσοκομείο της ΡΕΝ και άλλοι διακομίστηκαν με πολύ σοβαρά προβλήματα. Το πρόβλημα γύρω από αυτόν τον θάνατο είναι το εξής ότι δεν έχουμε να κάνουμε με διαφάνεια, αλλά με αδιαφάνεια όταν ένα εργαστήριο όπως το πορτογαλικό Μπιάλ δοκιμάζει κάποια μόρια. Το σχετικό πρωτόκολλο δημοσιεύθηκε στις 22 Ιανουαρίου στην Γαλλία, όμως δύο φακέλους δεν τους πήραμε. Ο ένας αφορούσε το πειραματικό φάρμακο που αφορούσε τις επιπτώσεις του ίδιου του φαρμάκου και δεν είδαμε και τις προκλινικές δοκιμές σε χιμπαζίδες εν προκειμένου. Αυτά δεν δημοσιεύθηκαν από τον οργανισμό και δεν μπορέσαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε πρόσβαση στους δύο φακέλους. Το πορτογαλικό εργαστήριο οχυρώνεται πίσω από το εμπορικό μυστικό. Η Κομισιόν και εσείς κύριε Επίτροπε μπορείτε να πιέσετε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να αποκτήσει πρόσβαση, και το που κυρία αυτό, στους φακέλους αυτούς. Αλλιώς θα πάμε στο 2018. Τότε θα δημοσιευθεί η σχετική βάση δεδομένων. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να πιέσετε να γίνει αυτό γρήγορα σήμερα. Να δημοσιευθεί αυτή η βάση δεδομένων για να αποκτήσουμε επιτέλους πρόσβαση στα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πεντητσίνη. Ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια μιας μελέτης φάσης 1 αξιολογούμε το φαρμακολογικό ε, προφίλ και την ανοχή των νέων μορίων. Γι' αυτό δεν εμπλέκονται πολλά άτομα. Πάντως πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε χρόνο έχουμε χιλιάδες θελοντές, συνήθως ε, νέους φοιτητές, που επειδή χρειάζονται κάποια χρήματα ε, συμμετέχουν σε αυτές τις κλινικές ε, δοκιμές ε, ρισκάροντας τη ζωή τους. Τώρα το κέντρο που έκανε την έρευνα και εδώ συμφωνώ πλήρως όμως είπε η συνάδελφος υπερασπίστε τον εαυτό του λέγεται ότι εφάρμοσε τους διεθνούς κανόνες και ακολούθησε πιστά όλε τι διαδικασίε. Εμεί όμω θέλουμε να ξέρουμε τι συνέβη πριν να φτάσουν στα πειράματα σε ανθρώπου, τι πειράματα έγιναν σε ζώα και ποιε άλλε δοκιμέ έγιναν πριν να τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινε ζωέ. Εμεί θέλουμε να ξέρουμε όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί. Γιατί ένα κλινικό θάνατο και ε, πέντε άνθρωποι με σοβαρέ επιπτώσει ε, είναι ε, πολύ ισχυρό πλήγμα και από ό,τι βλέπουμε πάρα πολλοί άνθρωποι σιωπούν για το τι συμβαίνει στον τομέα της υγείας. Πρόεδρος και τώρα, η κυρία Γκρουστέτ. Ευχαριστώ. Είναι αλήθεια ότι ε, ο θάνατος ενός εθελοντή είναι ένα δραματικό ατύχημα και φυσικά στέλνουμε τα συλληπιτήριά μας και στην οικογένειά του αλλά και στις οικογένειες των ανθρώπων που νοσηλεύονται. Άκουσα ότι το Υπουργείο Γαλλία, στην Γαλλία, το Υπουργείο Υγείας ζήτησε τη διεξαγωγή ερευνών για να διευκρινίσει το πώς έγινε αυτό το δράμα. Τώρα έχουμε πάρα πολύ μερικά στοιχεία για την υπόθεση αυτή. Συνεχίζονται οι έρευνες, επομένως ε, δεν θα πρέπει να κάνουμε εικασίες. Ε, δεν ε, ξέρουμε που είναι το λάθος στο πρωτόκολλο, ε, στο περιεχόμενο του δείγματος, στη δόση, στη χημική ουσία. Μπορούμε να φανταστούμε τα πάντα. Εδώ χρειαζόμαστε διαφάνεια. Όμως αυτό που πρέπει να επενθυμίσουμε είναι ότι οι κλινικές δοκιμές είναι απολύτως απαραίτητες για να θέσουμε στην αγορά καινοτόμα φάρμακα χρήσιμα στους ασθενείς και τέτοια ατυχήματα ευτυχώς είναι σπανιότατα και ευτυχώς ε, μας το υπενθύμησε και ο Επίτροπος, έχουμε ένα νέο κανονισμό που θα προβλέπει ισχυρές υποχρεώσεις διαφάνειας, κυρίως ό,τι αφορά ε, τις πληροφορίες για ε, τις δοκιμές στη φάση Α και την δημοσιοποίησή τους. Πρόκειται για απόλυτη προτεραιότητα, είναι σημαντικό και γι' αυτό απευθύνομαι στην Κομισιόν και στον ΕΟΦ να παρακολουθήσει την εξέλιξη αυτού του φακέλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Παρνιό. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, το δράμα, η τραγωδία της ΡΕΝ μας κάνει να αναρωτιόμαστε για πολλά ζητήματα. Καταρχάς, οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ε, έλαβαν γνώση ε, τέσσερις μέρες μετά για αυτές τις δοκιμές που έγιναν εξ ονόματος ενός πορτογαλικού εργαστηρίου. Νομίζω ότι αυτό αυτά τα εγγραφά που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση πρέπει να γίνουν δημόσια για να μπορούμε να γνωρίζουμε στην ουσία τι γίνεται σε τέτοιες δοκιμές. Με τους κανόνες που έχουμε από το 2014 ε, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ε, πληροφορίες για αυτές ε, τις δοκιμές και να γνωρίζουμε ποια είναι τα στάδια πριν δοθεί η έγκριση. Οι φαρμακευτικές εταιρείες όμως προσπαθούν να κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτό τον κανονισμό και την ισχύ του που θα τεθεί σε ισχύ το 2016. Υπάρχει μία διαδικασία η οποία επιτρέπει στις εταιρείες ε, να κάνουν λογοκρισία στις εκθέσεις ε, και να μην δίνονται τα στοιχεία που πρέπει ε, για αυτές τις κλινικές δοκιμές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει πλήρης δημοσιοποίηση των όλων των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με τις δοκιμές αυτές για να μπορούμε να είμαστε ε, να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Ε, θα πρέπει λοιπόν μετά από το ατύχημα στο ΙΡΕΝ να, έχουμε, να αναλάβουμε δράση έτσι ώστε ακόμα και για τέτοιες ε, δοκιμασίες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν μικρές επιπτώσεις να δίνονται τα στοιχεία γιατί δεν θέλουμε να έχουμε άλλον ένα σκάνδαλο στο τομέα της υγείας ε, ε, η Κομισιόν ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη της και αυτό το στοιχείο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ρίτσα, έχει ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ως φα... φαρμακολόγος που έχω λάβει μέρος σε κλινικές δοκιμές σε εμπορικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Ξέρω ε, πόσο ε, μεγάλη είναι αυτή η διαδικασία και πόσο δύσκολη. Κάποια από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα, όπως η ασπιρίνη για παράδειγμα, βάσει της διαδικασίας αυτής ε, δεν θα είχαν ποτέ λαβεί έγκριση. Σύμφωνα με την εμπειρία μου, τα αποτελέσματα ως τώρα, ε, ε, βάσει ας πούμε της ε, οδηγίας του 2001, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαδικασίες ήταν τόσο δύσκολες που τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου καλά. Και υπήρξε έτσι η παρεμπόδιση της έρευνας. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός που θα έχει πλήρη ισχύ φέτος θα είναι βελτίωση. Αμφιβάλλω όσον αφορά την αδιαφάνεια, Υποστηρίζουμε στο UKIP αυτή τη διαφάνεια. Θεωρούμε όμως ότι το Κοινοβούλιο και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ότι το Κοινοβούλιο είναι αυτό που θα πρέπει να ρυθμίζει αυτή τη διαδικασία και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ο κύριος Φερνάνετες έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, Κατερχήν ε, θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτεριά μου στην οικογένεια του θύματος και να ευχηθώ και περαστικά στους άλλους πέντε ανθρώπους που νοσηλεύονται. Οι εθελοντές που συμμετέχουν σε μια κλινική δοκιμή ξέρουν ότι διατρέχουν κινδύνους, όμως αυτοί οι κινδύνοι θα πρέπει να ελεγχιστοποιηθούν, να ελεγχθούν και να είναι ανάλογη με την σημασία των δοκιμών αυτών. Σε αυτό το περιστατικό που συζητάμε, αυτό που συνέβη ε, στην Γαλλία, ένας κατέληξε και πέντε είχαν ε, σοβαρές ε, συνέπειες. Πρέπει να γίνει διαφανής έρευνα, να βρούμε τις αιτίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, για να βρούμε τις αιτίες, χρειάζεται είναι θεμελιώδες ε, να γνωστοποιηθεί η αυτοψία αλλά και οι ιατρικές εκθέσεις τους ενδιαφερομένους και ε, με τις εκθέσεις αυτές θα μπορέσουμε να δούμε ποιες είναι οι αιτίες αυτού του ατυχήματος. Υπάρχει ε, επίσης ταχύς ρυθμός σε όλη την έρευνα. Βέβαια τίποτα δεν μπορεί να αποκρυφθεί, όλα θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν οι αιτίες. Και θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο αν οι ιατρικές εκθέσεις και η έκθεση της αυτοψίας έχει γνωστοποιηθεί, τουλάχιστον ε, αν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ πολύ. κύριος η κυρία Καμπεσόν Ρουίς, ευχαριστώ. Οι κλινικές δοκιμές είναι ουσιαστικέ ε, για να δοκιμάσουμε την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμάκων ε, και γι' αυτό πρέπει να συμμετέχουν οι ασθενείς, οι οποίοι πρέπει να είναι σίγουροι ότι τους εγγυόμαστε την ασφαλειά τους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την διαφάνεια. Ε, σίγουρα δεν είναι συνήθι γεγονότα στη Γαλλία, αλλά επίσης αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τα δεδομένα, δεν γνωρίζουμε τι συνέβη. Και φυσικά, όπως είπαμε αυτό, δεν μπορεί να παραμείνει κρυφό. Εδώ δεν είναι ε, η μόνη ε, διένεξη συμφερόντων που έχουμε και μας δείχνει την αναγκαιότητα αυτού του νέου κανονισμού. Αλλά νομίζω ότι χρειάζονται και νέα μέτρα για να βελτιώσουμε την απαραίτητη διαφάνεια υπέρ της ασφάλειας των ασθενών και για να προωθήσουμε και να βελτιώσουμε αυτή την έρευνα που είναι τόσο απαραίτητη για την αντιμετώπιση των νόσων. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζωρίνιο έχουμε, το πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο ε, και ταυτόχρονα να έχουμε ασφαλή φάρμακα. Αυτό είναι το ε, ερώτημα κλειδί για τους πολίτες και για την ε, δημόσια υγεία. Αυτό συζητούμε αυτή τη στιγμή. Η επιστημονική πρόοδος πρέπει να μας επιτρέψει να ε, σώσουμε χιλιάδες ζωές και να κατεπολεμήσουμε τις ε, νόσες. Όμως ε, χρειαζόμαστε διαφανή και ισχυρή νομοθεσία. Η απάντηση δεν είναι να έχουμε μια βαριά νομοθεσία, αλλά πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη διάδοση των γνώσεων και όπως είδαμε αυτά που έγιναν στη Γαλλία θα πρέπει να μας δώσουν περισσότερα κίνητρα προς την οδό που ακολουθούμε έχουμε την υποχρέωση να συνεργαστούμε περισσότερο και να συστήσουμε μια επιστημονική πλατφόρμα που να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που συνδέονται με τις κλινικές δοκιμές. Και γι' αυτό κύριε Επίτροπε σας συγχαίρω για την απόφαση να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων που θα υποστηρίζει όλη αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια των κλινικών ε, η ασφάλεια των ασθενειών ε, προστατεύεται με κάθε προσπάθεια όμως η τραγωδία της Γαλλίας μας δείχνει ότι δεν ισχύει πάντοτε ο θάνατος του θελοντή και τα πέντε άτομα που νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ε, ανάπτυξη ενό φαρμάκου είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι κάτι σπάνιο, όμως σε θέματα ασφάλειας ε, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Ο κανονισμός του 2014 για τις κλινικές δοκιμές θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο το 2018. Εν τω μεταξύ δεν μπορούμε να επιτρέψουμε άλλε τραγωδίες. Ο κανονισμός προβλέπει την αναγκαιότητα εις μελετών για να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν να χορηγηθεί ένα φάρμακο σε ανθρώπους και πρέπει να υπάρχουν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες πρέπει να δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία της φάσης 1 των πειραμάτων εμείς θα πρέπει να δούμε ποια είναι και τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για να προβούμε σε όσο δυνατόν ταχύτερη θέση σε ισχύ του κανονισμού. Ο τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο είναι η κυρία Λαουριστίν. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, και εγώ στέλνω τα συλληπιτήριά μου στα θύματα του τραγικού περιστατικού Κατανοούμε όλοι ότι αυτά αποδεικνύουν ότι η ψήφιση του κανονισμού τον Απρίλιο του 2014 πρέπει να ακολουθεί από εφαρμογή του. Θυμίζω μάλιστα ότι η πρώτη φάση δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό αυτόν. Εδώ τώρα μιλούμε για την βάση δεδομένων Και τι θέλουμε. Ε, αν πάμε στον Σεπτέμβριο του 2014, το είπε ο Επίτροπος, υποτίθεται ότι όλα θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, γιατί έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα μας πείτε λίγο περισσότερα για τη βάση δεδομένων. Τι θα περιλαμβάνει. Ωραία, πρόσβαση αλλά και θέλω μια εξήγηση, επαναλαμβάνω. Γιατί έχουν καθυστερήσει όλα αυτά τόσο πολύ, Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό ήταν και ο τελευταίος μιλητής εκ του καταλόγου. Κάτσου διάει, κύριε Σπότσακ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Είμαι πεπισμένος ότι δεν επιτρέπεται κλινικές δοκιμές να καταλήγουν σε θύματα νεκρούς ή στο νοσοκομείο. Πιστεύω ότι τα συμπεράσματα αυτής της ε, συζήτησης πρέπει να οδηγήσουν σε μια καλύτερη κατάσταση. Έλαβα τον λόγο για να υποστρίξω και τον Επίτροπο, ο οποίος ε, τάχθηκε υπέρ της αντικειμενικής πληροφόρησης. Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να συμβεί είναι ένας ε, αγώνας δρόμου που θα οδηγήσει σε ελληματική ενημέρωση. Αυτά ευχαριστώ για τη διαφάνεια και τον έλεγχο στη διαδικασία των κλινικών δοκιμών με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό στη γαλλία όπου είχαμε ένα νεκρό και πέντε άτομα τα οποία ακόμη κινδυνεύουν. οι κλινικές δοκιμές έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη των φαρμάκων και τη βελτίωση των φαρμακευτικών αγωγών που εφαρμόζονται ενώ εντός της ευρωπαϊκής ένωσης οι επενδύσεις στην κλινική έρευνα υπερβαίνουν τα είκοσι δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως ωστόσο συχνά παρατηρούνται περιπτώσεις έλλειψης διαφάνειας και ελέγχου στις κλινικές δοκιμές. επιπλέον συχνά παρατηρούνται περιπτώσεις απόκρυψης τυχόν αρνητικών αποτελεσμάτων στις προκαταρκτικές κλινικές δοκιμές και δημοσίευση μόνο των επιθυμητών αποτελεσμάτων επομένως προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια στις κλινικές δοκιμές θα πρέπει όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες να δηλώνουν και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα από τα πρώτα στάδια των κλινικών δοκιμών όπως άλλωστε ορίζει και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται τις αρχές δημόσιας υγείας, τις επιτροπές δοντολογίας και τις οντότητες που ερευνούν την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην αλήθεια και στη διαφάνεια. Θα πρέπει τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα σε σχέση με τα νέα φάρμακα που είναι υποδοκιμή και να είναι δημόσια και να μπορούν να μελετηθούν όπως πρέπει. Θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν δημοσιεύονται ε, οι μελέτες και οι γνωμοδοτήσεις των οργανισμών φαρμάκων αλλά και οι μελέτες των εταιριών που κάνουν κλινικές δοκιμές έτσι ώστε να ε, μπορούμε να σεβαστούμε και τις βελτίες πρακτικές. Χρειάζονται πληροφορίες για το πώς προχωρούν οι έρευνες και για τα ενδεχόμενα λάθη που έχουν ε, διαπραχθεί. Κανένα εμπορικό απόρριτο δεν μπορεί να αρνηθεί το δικαίωμα στην αλήθεια και στη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ. ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τα τραγικά γεγονότα στην Γαλλία. Μπορώ να πω ότι διαφάνεια είναι κάτι πολύ σημαντικό και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Επίτροπος. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καταρχάς να πω ξεκάθαρα ότι είναι ουσιώδης η διαφάνεια στις κλινικές δοκιμές είναι, ε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δοκιμές που διεξάγονται, πότε, από ποιον, ποιος είναι ο στόχος ε, και ποια τα αποτελέσματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε στενή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα πρέπει να έχουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες γιατί υπάρχουν προβλήματα σχετικά με τεχνικά ζητήματα αυτή τη στιγμή όσον αφορά στα δεδομένα. Μιλώντας τώρα για αυτό το τραγικό γεγονός στη Γαλλία, να πω ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες και από την γαλλική αστυνομία και από τις αρχές. Όμως ε, ε, τα αίτια δεν είναι ακόμα γνωστά. Υπάρχουν πολλές κλινικές υποθέσεις, ε, όμως δεν μπορούμε να σχολιάσουμε από νομική άποψη, δεν μας επιτρέπεται να σχολιάσουμε ε, τις έρευνες σε αυτό το στάδιο, γιατί είναι πολύ ευαίσθητη η κατάσταση. Πιστεύω ότι σύντομα θα γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Όμως πρέπει να ελέγξουμε πολύ καλά και να σας δώσουμε πληροφορίες όταν ολοκληρωθεί η έρευνα. Τότε θα μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήματα για τη διαφάνεια, για τις πληροφορίες. Όσο όμως τρέχουν οι έρευνες, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στοιχεία. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε, για τις διαβεβαιώσεις σας. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού